το Κοινοβούλιο να αποφανθεί και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο όσο γίνεται. Ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρίαση, λέει ο Ε, αύριο το πρωί επόμενη συνεδρίαση από τις 9 μέχρι τη 1 και το απόγευμα από τι 3 μέχρι τι 10 το βράδυ. Θα βρείτε την ημερήσια διάταξη και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Λίγη τη συνεδρίαση και σα ευχαριστώ πολύ.